την ισότιμη και δίκαιη και τίμια αντιπαράθεση. Και προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία από εδώ και μπρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, για τις εκλογές που θα γίνουν προς το θέμα των αντιπροέδρων. Θα πρότεινα μέχρι τις 6 και 30 το βράδυ να οριστεί η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ορίζεται αυτό ως προθεσμία. Και στο R00101 που ονομάζεται σημείο Προεδρίας, η Πασαρέλα Προεδρίας στο κτίριο που βρισκόμαστε, στο Λουίς Βάις, R00.101 και όχι 7 όπως είχε γραφτεί πριν. Ε, θα κατεθούν οι υποψηφιότητες μέχρι τις 6.30 στην Espace de la Présidence όπως ονομάζεται. Διακόπτουμε τώρα για να συνεχίσουμε στις 7.30 το βράδυ την συνεδρίαση της Συνόδου Λομελίας.